Ε, Διεθνούς Συνέλευσης της Δημοκρατίας της ε, Κορέας. Μόλις ήρθαν, βρίσκονται στα θεωρία, στα θεωρία των επισήμων. Όπως γνωρίζετε, η Δημοκρατία της Κορίας είναι πλέον ένας ε, στρατηγικός εταίρος προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πολλές κοινέ αξίες και αρχές και ε, προσπαθούμε να επιτύχουμε μαζί πολλές παγκόσμιες προκλήσεις. Έχουμε υπογράψει και μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου ιδιαίτερα ευρεία, η οποία ε, τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2011 και είναι και η πρώτη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου που απαιτούσε και υπογραφή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει των νέων κανόνων που καθορίζουν οι συνθήκες. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τους φίλους μας εδώ και θα έχω και την ευκαιρία να ε, προεδρεύσω στο κοινό γεύμα και να μοιραστούμε και κάποιες ε, σκέψεις και παρατηρήσεις για την κατάσταση στη χώρα τους, ε, για την κατάσταση της Κορεατικής Χερσονήσου και για τα όσα ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις ευρωεκλογέ ε, που προβλέπονται για το τέλος Μαΐου. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τους ε, φίλους και συναδέλφους από την Κορέα. Στο πρώτο σημείο που έχουμε στην ημερήσια διάταξη για σήμερα το απόγευμα... que hay una cuestión de orden ένα θέμα επί της διαδικασίας, δεν ξέρω από ποιον συνάδελφο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα, αλλά θα ήθελα απλώ να επισημάνω ότι δεν λειτουργούν τα ακουστικά μου και θα ήθελα να ζητήσω να έρθει ένας τεχνικός. Ευχαριστώ. Θα σας στείλουμε ένα τεχνικό για να μπορείτε να ακούτε και να μπορέσετε να παρακολουθήσετε και την υπόλοιπη συζήτηση της Ολομέλειας. Καταρχάς λοιπόν έχουμε τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής